Einen schönen Nachmittag für alle. Ich würde einfach mal anfangen wollen und bitte alle auf die Plätze zu gehen. Und Ας ξεκινήσουμε. Ε, να σας καλέσω όλους ε, να καθίσετε και να ακούσετε με προσοχή τα όσα θα σας πω. Η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται. Γι' αυτό δεν είναι πολύ καλό να ακούγονται ομιλίες. Λοιπόν, γνωρίζετε όλη την πρόταση της σημερινής ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω εάν υπάρχουν παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, τροποποίησεις, όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνεται. Όπως ήδη είπα, η σημερινή συνεδρίαση μεταδίδεται στο web stream. Και όπως πάντα, ελέγχουμε εάν χρησιμοποιούνται όλες οι καμπίνες διαρμηνίας και μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιούμε όλες τις γλώσσες, όλες τις καμπίνες της διαμηνίας λέει η Πρόεδρος. Η Επιτροπή Γυναικών μαζί με την Επιτροπή μας θα οργανώσει ακρόαση ε, σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων στις 19 Μαρτίου από τις 4 έως τις 6.30 το απόγευμα σχέδιο της ημερήσιας διάταξης θα σας σταλεί. Και μάλιστα είσαστε όλοι προσκεκλημένοι, όχι μόνο οι γυναίκες και οι άντρες να συμμετάσχετε. Έχω μία ανακοίνωση του κυρίου Ρή και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα προς ε, την Προεδρία της Επιτροπής μας. Γιατί η Επιτροπή μας ε, απάντησε στα ερωτήματά μας ε, σε ό,τι αφορά το Ταμείο για τους πλέον αδυνάμους. Υπήρχαν κάποια προβλήματα, κάποια ζητήματα σχετικά με τα social groceries και θα ήθελα να μας πείτε εάν έχουμε λάβει απάντηση της Επιτροπής σχετικά με τα social groceries και αν ναι, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι ακριβώς αυτή η απάντηση. Αυτά ήθελα να πω. Μας απάντησε με επιστολή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Έχουμε εδώ ένα τεχνικό πρόβλημα. Πάτσα λάθος κουμπί, δικό μου το φταίξιμο, λέει η πρόεδρο. Δυστυχώ δεν μπορώ να σας δώσω ικανοποιητική απάντηση. Θα μιλήσω όμως με την Περβάνς Μπερές. Αύριο θα είναι παρούσα, οπότε ελπίζω αύριο να μας απαντήσει. Λίγες ώρες υπομονή. Ελπίζω αύριο να έχουμε ικανοποιητική απάντηση σχετικά με τα ε, κοινωνικά παντοπολία. Ε, με ενδιαφέρει και εμένα το θέμα, άλλωστε. Ωραία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μία ερώτηση. Αναφερθήκατε σε διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή μας και μια άλλη Επιτροπή ε, αναφέρατε την 9η Μαρτίου που είναι Κυριακή. Επαναλαμβάνω λέει η Πρόεδρος. 19 Μαρτίου 4 με 6.30. Εντάξει. Και ούτως ή άλλως ε, θα σας σταλεί γραπτός η ενημέρωση. Σύντομα. Ώστε να μπορέσετε να προγραμματίσετε τη ζωή σας. Καλό θα είναι να εκπροσωπείτε και η Επιτροπή Απασχόλησης, διότι είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας πάρα πολύ. Κοιτώ τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Μέχρι τώρα δεν έχω λάβει καμία γραπτή παρατήρηση. Ούτε και εδώ βλέπω να υπάρχει καμία παρατήρηση. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Και προχωράμε στο πρώτο ουσιώδες θέμα της ημερήσιας διάταξης. και πρόκειται για τα δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. Η κυρία Όμεν Ρόιτεν είναι η συγγήτρια. Στις 4 Δεκεμβρίου η Κορεπέρ ενέκρινε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και η δική μας Επιτροπή ε, το Δεκέμβριο ενέκρινε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Και τώρα το θέμα είναι ότι και το Συμβούλιο θα εγκρίνει το αποτέλεσμα. Υπάρχουν ακόμα τα τεχνικά ζητήματα, το θέμα το γλωσσικό. Όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά, μπορεί να πάει το θέμα στην Ολομέλεια και εντό στις θητείες μας να εγκρίνουμε το ε, θέμα αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι αλλιώς ε, χάνουν οι ε, μετακινούμενοι εργάτες τα δικαιώματα αυτά. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτριά μας, την κυρία Όμεν Ρόιτεν. 17 Δεκεμβρίου είπε η Πρόεδρος, νομίζω ότι εγκρίνει το Συμβούλιο, μετά θα πάει στην δεύτερη ανάγνωση. 17 Φεβρουαρίου, λέει η Πρόεδρος, ε, θα αποφασίσει το Συμβούλιο, κατόπιν ε, θα διαβιβαστεί σε εμά το θέμα και υποθέτουμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο θα συζητηθεί το θέμα, δηλαδή 18 Μαρτίου εδώ θα συζητηθεί το θέμα και στην τελευταία συνεδρίαση του Απριλίου θα γίνει ψηφοφορία. Υπάρχουν παρατηρήσεις, όχι, ωραία, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η ενδιάμεση έκθεση του κυρίου Έρι σχετικά με απόφαση του συμβολίου για την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Δίνω το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Ήρη. Eh, eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ε, πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολη περίπλοκη έκθεση, όμως ε, είναι μια σημαντική ε, έκθεση για όσους ε, τους απασχολεί αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής. Πρόκειται για μια σύνοδο κορυφής ε, που διοργανώνεται πάντα στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής και μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων. Μιλάμε λοιπόν για μια τριμερή κοινωνική σύνοδο που διαθέτει νομική βάση και το νομικό της πλαίσιο έχει τροποποιηθεί ελαφρώς εξαιτία των νέων κανόνων που δημιουργήθηκαν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τα εξήγησα όλα την προηγούμενη φορά, μιλήσαμε με εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου και σήμερα μάλιστα συνομίλησα με εκπροσώπους ε, των σωματείων. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά υπήρξαν διαβουλεύσεις με όλους, γνωρίζω τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών. Βεβαίως ε, και τα λόμπι προσπάθησαν να ασκήσουν πίεση, αφενός από ε, την πλευρά των εργαζομένων και από την, αφετέρου από την πλευρά των εργοδοτών. Υπάρχουν σωματεία που θα ήθελαν ε, μεγαλύτερη επιρροή σε αυτή τη διαδικασία όχι μόνο ως ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας ε, Σωματείων, αλλά και ως ε, μεμονωμένα συνδικάτα. Είχαμε λοιπόν κάποιες επαφές από πλευρά εργαζομένων και εργοδοτών. Chambers. Σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς εταίρους, έχουν ήδη δικές τους δομές και σύστημα Επομένω, ε, εφόσον έχουμε ήδη το πρωτόκολλό μας και δεν έχουμε και τόσο μεγάλο χρονικό περιθώριο, θα μείνουμε εκεί. Εγώ μίλησα για αυτό το ζήτημα, ανέφερα αυτό το ζήτημα και στις τροπολογίες. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι ακόμα και η Business Europe αλλά και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ε, Σωματείων και Συνδικάτων θα πρέπει να μεταφέρουν τις απόψεις τους ε, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Πρέπει λοιπόν ε, να ακουστεί και η γνώμη των ε, συνδικάτων και των εργαζομένων. Δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, όμως πρόκειται για μια υποχρέωση πλέον να περάσουμε, να διαβιβάσουμε όλες τις απόψεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι συμφώνησαν <coughs> οτιδήποτε αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής να είναι μόνο μια αποκριστάλλωση των όσων κάναμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε για υφιστάμενες πρακτικές. Για τις τροπολογίες, τώρα έχουμε δύο συμβιβαστικέ, την Α και τη Β. Η Α αφορά του ε, σοσιαλιστές ε, και την ΑΛΔΕ. Παντρέψαμε δύο τροπολογίες ουσιαστικά. Νομίζω ότι οι οικολόγοι, οι σοσιαλιστές και το ΕΛΚ θα συμφωνήσουν σε ό,τι αφορά αυτή την πρώτη ε, συμβαστική. Για την Β υπάρχει ένα νέο στοιχείο. Υπάρχει μια ε, διαφορά απόψεων μεταξύ του ΕΛΚ και των ε, σοσιαλιστών σε ό,τι αφορά το ρόλο του Κοινοβουλίου. Αν θα έχει το Κοινοβούλιο το δικαίωμα να συμμετάσχει ε, σε αυτή την ε, Σύνοδο Κορυφής. Κατά τη γνώμη των σοσιαλιστών θα πρέπει να στείλουμε μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στην κοινωνική συνοδοκορυφή. Όμω ούτε οι εργοδότε ούτε οι εργαζόμενοι συμφωνούν με αυτή την πρόταση. Γιατί είναι λίγος ο χρόνος και γι' αυτό θα ήθελαν να αξιοποιήσουν αυτό το χρονικό διάστημα με καλύτερο τρόπο. Οι σοσιαλιστές λοιπόν δεν συμφωνούν με μας Ποιοι θα παρίστανται σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, ε, Υπουργός ε, της ε, Ελληνικής Προεδρίας αλλά και των επερχόμενων Προεδριών, πολύ καλά όλα αυτά, όμως νομίζω ότι πάνω απ' όλα πρόκειται για έναν διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Δεν είναι λοιπόν απαραίτητο να στείλουμε μια ολόκληρη κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να στείλουμε κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία γιατί πρόκειται για κοινωνικό διάλογο, διάλογο μεταξύ κοινωνικών εταίρων. Και αν οι εργαδότες και οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να προσκαλέσουν απαραίτητα μία ε, κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία δεν πρέπει να το ε, πιέσουμε παραπάνω γιατί δική του είναι η συνόδος κορυφής δικός τους είναι ο διάλογος, αυτοί αποφασίζουν. Αυτές λοιπόν είναι οι θέσεις ε, των σοσιαλιστών λοιπόν μιλούν για μια υποχρεωτική παρουσία κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία με την οποία πρόταση εγώ δεν συμφωνώ. Σα εξήγησα ήδη γιατί η κοινωνική αυτή τη σύνοδο κορυφή δεν είναι δική μα. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τον διάλογό του με αυτή την κοινωνική σύνοδο που οργανώνουν. Αυτοί θα αποφασίσουν ποιου θέλουν να προσκαλέσουν και ποιου όχι. Δεν μπορούμε να τους αναγκάσουμε να προσκαλέσουν ε, ε, μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία. Βεβαίω η συμμετοχή σε μια τέτοια σύνοδο κορυφή ε, έχει τα πλεονεκτήματά τη για μα. Θα ήταν καλό να δούμε πώ ακριβώ διεξάγεται αυτή η σύνοδο κορυφή. Όμω, επαναλαμβάνω, πάνω απ' όλα είναι σύνοδο κορυφή των κοινωνικών εταίρων. Δεν συμφωνώ με τι τροπολογίε Μπέκερ. που κάνει λόγο για εκπροσώπηση των ε, εργοδοτών και των εργαζομένων. Δεν νομίζω ότι είναι δικός μας ε, ρόλος να αποφασίσουμε πόσοι εκπρόσωποι των εργοδοτών και πόσοι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα συμμετάσχουν. Εκείνοι θα αποφασίσουν μόνοι τους, έχουν τις δικές τους δομές και διαδικασίες που λειτουργούν μια χαρά. Δεν συμφωνώ λοιπόν με την τροπολογία Μπέκερ. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Δεν θα υπάρξουν λοιπόν προβλήματα αύριο στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Yeah. Vielen Dank, äh, lieber Kollege. Ναι, αγαπητέ συνάδελφε ε, Ρή, ευχαριστώ πολύ. Είναι σειρά τώρα των σκιωδών εισηγητών και από το SND. Είναι η συνάδελφος ε, Μπαλταχίνο, παρακαλώ. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καταρχήν προωθήσαμε το θέμα της ε, συνεργασίας για αυτό το ζήτημα. Σήμερα το πρωί είχαμε μια ιδιαίτερα επικοδομητική συνάντηση με τα συνδικάτα και Επίσης ενημερωθήκαμε για την ανάγκη και το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη δημιουργία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που μόλις προείπε ο κύριος Ορή που αφορά το ε, καθεστώς του παρατηρητή που ζητούμε. Ελπίζουμε δηλαδή να λάβουμε αυτό το καθεστώς του παρατηρητή σε αυτή τη διάσκεψη κορυφής. Αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα σε αυτή την τροπολογία συμβιβασμού έτσι ώστε η Επιτροπή Απασχόλησης να λάβει αυτό το καθεστώς παρατηρητή. Την προηγούμενη εβδομάδα το συζητήσαμε, αλλά φαίνεται ότι αλλάζουμε θέση. Το συζητήσαμε, όπως σας είπα, το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κατάρτιση των ευρωπαϊκών πολιτικών και επειδή έχουμε ευθύνη για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές θα πρέπει να λάβουμε αυτό το καθεστώς του παρατηρητή στη διάσκεψη κορυφής του καλοκαιριού. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν την χάνει υποστήριξης, δηλαδή να μιλήσουμε για την δυνατότητα της Επιτροπής αυτό την, ε, τον τριμερή διάλογο να μπορέσει ε, να προωθηθεί μέσα στα πλαίσια της διάσκεψης κορυφής, ε, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων. Με βάση αυτές τις συζητήσεις ε, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό. Παρά να τα αποπέμψουμε. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο ούτε βλέπω την ε, σκιώδη συγγήτρια Χάρκιν. Α, και όμως. Όχι, δεν είναι παρούσα. Η Καρυματέλη δεν είναι παρούσα. Η κυρία Μάκεντάρ δεν είναι παρούσα. Οι σκιώδεις συζητητές φαίνεται ότι παρακολουθούν το θέμα από το γραφείο τους. Ε, Ε, γι' αυτό δίνω το λόγο στον Τόμας Μαν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι, πάντα είναι καλύτερο να είμαστε παρόντες. Ε, θα ήθελα να καλέσω τους σοσιαλδημοκράτες ε, να ε, κάνουμε ένα συμβιβασμό. είναι δύσκολο το θέμα. Σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε τονίσει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και αν καταλήξουμε σε αποτέλεσμα, ε, τότε ισχύει και το αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε παρόντες ως παρατηρητές. Εκ των υστέρων, θα ε, ακούσουμε την έκθεση αν είχαμε επιτυχία ή όχι και η Επιτροπή Απασχόλησης ε, σίγουρα θα λάβει υπόψη το θέμα αυτό. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε καθεστώς παρατηρητή. Έχω δει πολλές αντιπροσωπείες ε, να ε, σε συγκαλούνται με πολλή προσπάθεια, τελικά να μην είναι παρόν κανείς, ε, υποχρέωση λογοδοσίας δεν έχουν και συνεργαζόμαστε επί πολλές δεκαετίες. Συμφωνώ πολύ με τον Τσάπα Ούρι. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν το καθεστώς του παρατηρητή, άλλωστε θα ενημερωθούμε για το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θεωρούμε φίλους τους κοινωνικούς εταίρους, έχουμε καλές κοινέ παραδόσεις και δεν χρειαζόμαστε ε, κάτι τέτοιο. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ, καλή, πολύ καλός ο συνδεσμός του Τσάμπα Το ΕΛΚ και η ε, πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες ε, νομίζω τελικά θα καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα θα είναι ε, αυτό είναι ένα συμβασμό στον οποίο μπορούμε να δεχτούμε. Θα μιλήσω αγγλικά, λέει η Πρόεδρο. Ε, Μαριον Χάρκεν, μιλάμε για ε, την τριμερή διάσκεψη κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη διότι έφτασα αργά. Καταρχήν έχω μία ερώτηση προς την Επιτροπή. Διαβάζοντας το κείμενο, κοιτώ το συμβιβασμό Β και διαβάζοντας το κείμενο της Επιτροπής αναφέρει ότι ε, εξαρτώμενο από την ε, ημερήσια διάταξη και με βάση την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Προεδρίας και της Επιτροπής και ούτω καθεξής, από ό,τι καταλαβαίνω θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση, διότι αυτό σημαίνει η πρόταση αυτή. Και η ερώτηση είναι θα συμμετέχουν ως παρατηρητές ή θα συμμετέχουν στην συνάντηση κάθε αυτή. Έχουμε υποβάλει το ερώτημα και δεν έχουμε λάβει απάντηση. Ίσως αυτό θα μπορούσε να αποσαφινιστεί. Γιατί αν δείτε τη δική μας πρόταση συμβιβασμού για την τροπολογία Β, μιλάμε για την Προεδρία της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων που έχει προσκληθεί που σημαίνει ότι δεν θα έχουμε στάτους παρατηρητή, θα συμμετέχουμε στη συνάντηση. Για να διασαφίσουμε αυτό το ζήτημα θα ήθελα να ακούσω την Επιτροπή. Μέχρι τώρα δεν είναι σαφές. Πέρα από αυτό, η άποψή μου είναι εάν θεωρούμε ότι η Προεδρία, η Πρόεδρος θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία δεν πρέπει να εξαρτάται από την ημερήσια διάταξη, διότι η ατζέντα θα αφορά την ανεργία παγκοσμίως. Γι' αυτό ε, προβλέπεται και αυτή η κοινωνική διάσκεψη κορυφής. Θεωρώ ότι άλλοι υπουργοί από άλλα υπουργεία οικονομικών γεωργίας και ούτω καθεξής και άλλοι επίτροποι που δεν έχουν άμεση ευθύνη για θέματα απασχόλησης ε, και ανεργίας καθώς και κοινωνικής ανάπτυξης επειδή ε, η ατζέντα αφορά κοινωνικές υποθέσεις και ανάπτυξη, θεωρώ ότι, το, ότι η Προεδρία της Επιτροπής θα είναι παρούσα. Ελπίζω αυτό να είναι σαφές. Ναι, ευχαριστώ πολύ Μαριαν Χάρκιν. Σκοπεύουμε να καλέσουμε την Επιτροπή να απαντήσει σε κάποιες από τις ερωτήσεις και να μας ξεκαθαρίσει και τη διαδικασία. Με ενημέρωσαν ότι ο κύριος Ζαν Τρικά είναι παρόν. Όχι. Δεν είναι ο ίδιος παρόν, αλλά κάποιος άλλος. Από το τμήμα για τον κοινωνικό διάλογο και τις ε, σχέσεις ε, με τους οικονομικούς φορείς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι. Ε, είχα εδώ για να αντικαταστήσω τον συνάδελφο. Σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα που ετέθη, Εν συντομία θα ήθελα να σας πω ότι το καθεστώς του παρατηρητή δεν ε, υφίσταται, δεν αναφέρεται στην απόφαση που θεσπίζει αυτή τη σύνοδο κορυφής την τριμερή. Δεν υπάρχει καθεστώς παρατηρητή. Τώρα για τους εκπροσώπους των, ε, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν τμήμα της ε, αντιπροσωπείας των δύο αυτών θεσμικών οργάνων. Τα ίδια θεσμικά όργανα λοιπόν αποφασίζουν ποιο ε, θα συμμετάσχει στη συνοδοκορυφή. Ελπίζω να είναι σαφή τώρα τα πράγματα. Ähm, Ωραία. Θέλω ε, να θέσω μια συμπληρωματική ερώτηση. Αυτό δεν συνηθίζεται, αλλά μου φαίνεται απαραίτητο καθότι υπάρχουν κρεμότητες. Θα πρέπει αυτό να το καταλάβουμε ως εξής, ότι η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Και κύριε Ρή, έχετε κι εσείς κάποια ερώτηση ή θέλετε απλά να συνοψίσετε ούτως ή άλλως θα σας δώσω το λόγο μετά. Ε, εντάξει, θα σας δώσω το λόγο για να συνοψίσετε, αλλά θα παρακαλούσα την Επιτροπή να απαντήσει. Σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε σχετικά με τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντική για τη λήψη απόφασης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση της Επιτροπής υπευλήθη επί της νομικής βάσης ε, του άρθρου 351 του ιστορικού Κανονισμού και σε σχέση με κάποιες χώρες όπως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία ε, συμπεριλαμβάνεται μία εσωτερική έγκριση, κύρωση που παίρνει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει ε, μία και μόνο νομοθετική πράξη που προτείνεται κάθε χρόνο, bill στα αγγλικά, που συμπεριλαμβάνει όλες αυτές τις προτάσεις που βασίζονται στο άρθρο 351 της συνθήκης. Για το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες για να γίνει αυτό το ίδιο. Συμβαίνει και στη Γερμανία. Γι' αυτό αυτές οι δύο χώρες δεν μπορούν να κυρώσουν προς το παρόν το κείμενο. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον συγκεκριτή, τον κύριο Τσάπαουρη. Ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι η διαδικασία κύρωσης ε, διαφέρει μεταξύ κρατών μελών και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό προφανώς. Όμως ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια τεχνική και μόνο τροποποίηση. Ουσιαστικά πρέπει να θέσουμε επί χάρτου μια πρακτική που υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Είναι μόνο τυπική διαδικασία λοιπόν. Απλώς μεταφέρουμε στο κείμενο κάτι το οποίο ισχύει εδώ και καιρό. Μόνο αυτό συμβαίνει. Πράγματα που συμβαίνουν εδώ και πρακτικές που ισχύουν εδώ και χρόνια στην πράξη μεταφέρονται πλέον και στο κείμενο. Βεβαίως μεγάλες αλλαγές σίγουρα δεν θα γίνουν δεκτές ε, με ενθουσιασμό. Σε ό,τι αφορά τη δική μου τροπολογία, αν δείτε την τελευταία φράση, πρόταση, αναφέρει ότι σύμφωνα με την μέσα διάταξη, ανάλογα με την μέσα διάταξη, μπορούν να ε, προσκληθούν και άλλοι υπουργοί ή συμμετέχοντες. Μπορούμε ίσως να προσθέσουμε και τον, την πρόεδρο της ε, Επιτροπής Απασχόλησης του Κοινοβουλίου. Όμως, ας δώσουμε τον τελευταίο λόγο στους κοινωνικούς εταίρους. Να πούμε δηλαδή ότι μπορούν να προσκαλέσουν οι κοινωνικοί εταίροι εάν ε, το επιτρέπει ε, η μέρη στα διάταξη. Μπορούν λοιπόν να προσκαλέσουν αυτή την περίπτωση τον την πρόεδρο της ε, Επιτροπής Απασχόλησης γιατί αν είναι υποχρεωτική αυτή η πρόσκληση, τότε δεν πρόκειται πλέον για τριμερή σύνοδο αλλά τετραμερή. Δεν είναι αυτό ο στόχο μα. Έχουμε λοιπόν ε, κάποιες διαδικασίες για να μάθουμε σε μεταγενέστερο στάδιο τα αποτελέσματα αυτής της Συνόδου Κορυφής. Επομένως δεν χρειάζεται σώνη και καλά να συμμετάσχουμε. Και η ημερήσια διάταξη σίγουρα θα συνδέεται στενά και με την ημερήσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής. Τα ίδια ζητήματα θα τους απασχολήσουν. Δεν είναι λοιπόν και απαραίτητο να προσκληθούμε και ούτε χρειάζεται να είμαστε και βασιλικότεροι του βασιλέως, ας αφήσουμε σε αυτούς την απόφαση αυτή. Äh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κλείνουμε το, τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Αύριο είναι η ψηφοφορία και στην ε, Ολομέλεια του Μαρτίου θα είναι το θέμα στην ημερήσια διάταξη, από ό,τι μπορούμε να περιμένουμε. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Αύριο είναι η ψηφοφορία. Σήμερα μπορούμε να συζητήσουμε την γνωμοδότηση της Ιούτα Στάινρουκ σχετικά με την εσωτερική ναυσιπλοεία. Και την παρακαλώ πολύ σύντομα να μας παρουσιάσει το θέμα. Κατόπιν θα δώσω το λόγο στους κοιόδης συζητητές. Παρακαλώ, Γιούτα. Ευχαριστώ πολύ, Ελίζαπετ. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τους σκιώδεις συζητητές ε, για την ε, πολύ εντατική και επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Θα ήθελα να επανέλθω στις ε, συζητήσεις που είχαμε. Κατά τη διάρκεια της ε, συζήτησης στην επί της ουσίας σε αρμόδια επιτροπή. Με κατηγόρησαν ότι θέλω να δημιουργήσω ένα κοινωνικό ταμείο από ένα περιβαλλοντικό ταμείο. Θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση της Κομισιόν. Τα μέτρα καλύπτουν μόνο κοινωνικές πτυχές. Τα μέτρα αυτά μπορούν να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν και μέτρα εκπαίδευσης. Τη διοργάνωση του τομέα, καθώς και καινοτομία και καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση. Δεν δημιούργησα λοιπόν εγώ αυτό το ταμείο, αλλά στο πνεύμα του άρθρου 8 για το οποίο ε, είμαστε αρμόδιοι, το έχω επεξεργαστεί. Θα έχουμε λοιπόν ε, δύο συμβαστικές τροπολογίες. Τη συμβαστική τροπολογία Α σχετικά με, την, ε, με το δικαίωμα μετεκπαίδευσης και η Β που έχει να κάνει με τη βελτίωση της ικανότητας για τους ιδιοκτήτες αλλά και για τους εργαζομένους. βρίσκω πολύ κρίμα ότι και το ΕΛΚ και η ΑΛΤΕ δεν ήταν διατεθειμένοι να υποστηρίξουν περαιτέρω συμβιβαστικές τροπολογίες. Ακούσαμε για το θέμα των κοινωνικών εταίρων και για μένα ήταν σημαντική προϋπόθεση η πόροι να διατίθενται προς όφελος ε, το, της απασχόλησης στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Θέλω λοιπόν να υπάρχει συμμετοχή και των ε, ε, εργοδοτών και των εργαζομένων. Είναι και οι δύο κοινωνικοί εταίροι. Οι κοινωνικοί εταίροι γνωρίζουν τις ανάγκες, έχουν διαφορετική οπτική γωνία και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ καλό να υπάρξουν συνομιλίες. Ελπίζω πολύ σύντομα να έχω τη Ελπίζω σήμερα να έχω σύντομα τη δυνατότητα να αναφερθώ σε διάφορα θέματα που αφορούν τα επιμέρους άρθρα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα πω τα ονόματα των σχεδόν εισηγητών. Ο David Κάζα από το ΕΛΚ, δεν τον βλέπω. Α, η Τανούτα Γιασοψιέσκα έχει λάβει εντολές από τον David Κάζα, τη δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να, με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τον κύριο Στάινρουκ για την κυρία Στάινρουκ ε, τη κράτησε συμβαστική στάση κατά τις διαπραγματεύσεις. Θα υποστηρίξουμε τις τροπολογίες Α και Β. Όμως δεν θα υποστηρίξουμε άλλες τροπολογίες που αλλάζουν το πεδίο εφαρμογής. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην ε, τελική μας τάση. Ευχαριστούμε, Ντανούτα. Ωραία. Από ε, την Άλτε, ο Φίλιπ Τεπάκια δεν τον βλέπω. Αλλά ο Φίλιπ Πένιον έχει το λόγο, παρακαλώ. I'm speaking... Μιλώ εξ του Φίλιπ Μπάκερ θα ήθελα να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για την εργασία της διότι ε, οργάνωσε και συνεδριάσει σκιωδών όπου φτάσαμε σε δύο συμβασμούς. Η Επιτροπή έκανε μια καλή ε, πρόταση και θεωρεί όμως ότι δεν πρέπει να αλλάξει. Η Επιτροπή Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει ειδική χρήση των ταμείων. Οι πόροι όμως δεν είναι απεριόριστοι και θα, μας ενδε... θα πρέπει να μας ενδιαφέρει ε, το greening του στόλου. Μιλάμε για 35 εκατομμύρια ευρώ και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρησιμοποιούνται σε εσωτερικές φλωτές οδούς περίπου 10.000 μαούνες και προβλέπονται 3.500 ευρώ για κάθε μαούνα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους διαθέσιμους πόρους ε, προωθώντας την καινοτομία και δελεάζοντας τους νεότερους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ταμείο σαν ταμείο συνταξιοδότησης. Γι' αυτό θα πρέπει να συμφανίσουμε επί μιας πρότασης ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Έτσι θα προωθήσουμε τις εσωτερικές πλωτές οδούς για τη μεταφορά αγαθών έτσι ώστε να είναι μια αξιόπιστη εναλλακτική στις οδικές μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι σκιώδης για τους πράσινους. Δεν βλέπω κανένα άλλο. Εγώ λοιπόν μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Οι συμβαστικές προτάσεις έχουν τη μορφή που περίπου είχαμε φανταστεί, τουλάχιστον όσον αφορά τις δικές μας τροπολογίες. Ελπίζω αύριο να έχουμε επιτυχή ψηφοφορία. Αυτά από μένα και δίνω τώρα το λόγο στην Κομισιόν για το θέμα αυτό. Στον κύριο Θεοδολογίδη. Sie haben das Wort, bitte. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ. Πολύ καλά τα καταφέρατε με το όνομα. Θεολογίδης ονομάζομαι. Πράγματι, καταρχήν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για την ενδελεχή εργασία της που έγινε με μεγάλη σπουδή. Η Επιτροπή Τραν ε, το ίδιο, την ίδια στάση δείχνει καθώς και το Συμβούλιο και προωθούμε συζητήσεις έτσι ώστε να επέλθει συμφωνία ήδη κατά τη θητεία αυτή μέχρι τον Απρίλιο ή Μάρτιο ή Απρίλιο. Εκτιμούμε τις εργασίες σας, μπορούμε να υποστηρίξουμε όλες τις τροπολογίες που σχετίζονται με θέματα κλίματος, ε, περιβάλλοντος και καινοτομίας. Υποστηρίζουμε επίσης τις τροπολογίες οι οποίες σχετίζονται με πληροφόρηση και διάδοση πληροφοριών, αν και δεν θα πρέπει να αποτελέσουν υποχρεωτικό ενδιάμεσο στάδιο, γιατί όλα θα ε, τα περιμένετε από την Επιτροπή και μέχρι να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες δεν θα διαθέτετε τίποτα. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να είναι ένα μέσο διευκόλυνσης αλλά όχι πρόκριμα των μέτρων. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα των εσωτερικών πλωτών οδών, θεωρούμε ότι οι οικονομικοί φορείς αποτελούν ένα τόσο ευρύ πεδίο όπου μπορούν να συμπεριληφθούν και εκείνοι που δεν είχαν αρχικά συμμετάσχει. Άρα θα πρέπει να το διασαφίσουμε αυτό. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που μας βρίσκει σύμφωνους, όχι όμως με τον τρόπο που έχει παρουσιαστεί, αφορά την δημιουργία ενός κοινωνικού ταμείου όπου θα συμμετάσχουν και οι κοινωνικοί εταίροι. Αν και θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση ε, κινείται προς την κοινωνική πτυχή του ζητήματος, τι μας λέει αν μειωθεί η ικανότητα, δηλαδή εάν ο στόλος αποχωρήσει από την αγορά, τότε θα πρέπει να λάβετε ε, αντισταθμιστικά μέτρα για αυτούς τους ανθρώπους. Άρα η βάση είναι κοινωνική. Και αυτό έχει ενισχυθεί γιατί η αρχική πρόταση προέβλεπε μόνο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ότι οι ιδιοκτήτες δηλαδή θα ευεργετηθούν. Αλλά εμεί θεωρούμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα ευεργετηθούν. Αν βγει από την κυκλοφορία ε, ένα πλοίο, τότε θα ευεργετηθεί και ο καπετάνιος αλλά και τα μέλη του πληρώματος. Γιατί φοβόμαστε όταν μιλάμε για κοινωνικούς εταίρους. Ε, δεν είναι μυστικό ότι όταν ε, θέλουμε να φτάσουμε σε συμφωνία μεταξύ κοινωνικών εταίρων αυτό είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο εγώ έχω ασχοληθεί με το θέμα των ορών εργασίας και ανάπαυσης στις εσωτερικές πλωτές οδούς και χρειάστηκαν 7 χρόνια γι' αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάτε ότι αρχίσαμε το 2006 και φτάσαμε σε ένα συμπέρασμα στις αρχές του προηγούμενου έτους. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία. Εφόσον πρόκειται για πρόκριμα για να απελευθερώσουμε τα μικρά αυτά κονδύλια, του αποθεματικού, αυτό θα μπορούσε να δυσχεράνει τη διαδικασία, διότι το ταμείο αυτό συστάθηκε το 1999 και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Γι' αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει η διευκόλυνση της χρήσης, βασιζόμενη στο γεγονός ότι πρόκειται για μία πρόταση κοινωνικού προσανατολισμού και να μην δυσχεράνουμε το πλαίσιο λειτουργίας. Γι' αυτό θα θέλαμε να ε, λάβετε υπόψη αυτή την πτυχή κατά την αυριανή σας απόφαση. Σας ευχαριστώ και τέλος η συγκήτρια Ιούτα και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο ρόλος ε, των κοινωνικών εταίρων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί εταιρική σχέση ακριβώς και οι εμπειρίες από τα κράτη-μέλη μας δείχνουν ότι οι χώρες όπου οι κοινωνικοί εταίροι έχουν κοινό ρόλο, ε, έχουν και τη μεγαλύτερη επιτυχία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Κομισιόν με τον αποκλεισμό τους μάλλον περιπλέκει τα πράγματα. Μάλλον έχει διαφορετική όσον αφορά τη χρήση των πόρων. θα πρέπει να συνοδεύουμε, να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους, όχι μόνο τους ε, ιδιώτες, αλλά και τους ε, εργαζομένους ε, στα πλοία. Το ταμείο αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε και γι' αυτό τροποποιήθηκε το άρθρο 8, στο οποίο η Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να καλύπτει κοινωνικές πτυχές. Δεν νομίζω ότι το άρθρο 8 αυτό θα πρέπει να έχει σαν στόχο την οικολογικοποίηση της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αύριο. Νομίζω ότι θα είναι χαμένη ευκαιρία εάν δεν λάβουμε υπόψη μας και τους δύο κοινωνικούς εταίρους εδώ πέρα, διότι είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε έτσι να κλείσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Όπως ήδη ανέφερα, αύριο θα ψηφίσουμε. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών θα πραγματοποιηθεί 20 Φεβρουαρίου και στον Απρίλιο, κατά την τελευταία συνεδρίαση δηλαδή, θα πάει το θέμα στην Ολομέλεια, υπολογίζουμε. Διστάζω τώρα λίγο, διότι το επόμενο σημείο είναι η έκθεση του συναδέρφου Σέρκας και θα ήθελα πολύ να του δώσω το λόγο. Το θέμα είναι οι πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικας στις χώρες του προγράμματος της ζώνης του ευρώ. Μας ενδιαφέρουν εδώ οι κοινωνικές πτυχές. Παρακαλώ, κύριε Τσέρκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Η πρόεδρος ε, Περβάνς Μπερές ε, μου υποσχέθηκε να είναι ευρύτερη η συζήτηση από ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Δέκα λεπτά, δέκα λεπτά. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την γραμματεία της Επιτροπής αλλά και όλων των πολιτικών ομάδων διότι ήταν ευρύτατη η διαδικασία. Είχαμε 244 τροπολογίες και φτάσαμε σε 32 τροπολογίες συμβιβασμού. Ήταν πολύ ικανοποιητική η συνεργασία αλλά συζητήσαμε το ζήτημα με την κυρία Ρετζίνα Μπάστος εκτενώς και διανύσαμε ε, δύσκολες στιγμές από το 1385 από τη μάχη της Αλζουμπαρότα. Ξέρετε ότι οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί ε, αντιμάχονται οι τους δε. Και η, κυρία αυτή ήταν άξια συνεχιστής αυτής της ε, ε, μάχης που είναι γνωστή στην ιστορία μεταξύ των Ιβύρων. Εν πάση περιπτώσει καταφέραμε να συμφωνήσαμε, να συμφωνήσουμε, δεν συμπεριλάβαμε τροπολογίες που σχετίζονται με, την επιτροπή, με τις επιτροπές ΑΦΚΟ και ΕΚΟΝ. Και δεν ε, ασχοληθήκαμε με ζητήματα που δεν άπτονται των τεσσάρων χωρών, των χωρών που υπάγονται σε πρόγραμμα και που είχαν επιπτώσει στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων. Ε, εγώ στους συμβιβασμούς δεν ήθελα να ε, φτάσω σε εθνικές αντικσότητες, δηλαδή μιλήσαμε για τις χώρες αυτές μέσα στα πλαίσια μιας εγκαρσιότητας και ε, εγκάρσιων λύσεων, χωρίς να πούμε σε εθνικά ζητήματα. Είχαμε να κάνουμε όμως με δύο στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τους συμβασμούς και έχουν να κάνουν ε, με θέματα ευθύνης. Ε, εγώ ασχολήθηκα με θέματα τρόικας αποκλειστικά Μίλησα για μία κακή ε, οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση ε, η οποία έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Και επίσης ε, ασχοληθήκαμε με ζητήματα κατανομής ευθυνών μεταξύ Τρόικας και κρατών μελών. Πιστεύω ότι φτάσαμε σε μία εξισορρόπηση όπου γίνεται κατανομή ευθυνών με τις τροπολογίες α, β, γ και η και στο συμβασμό Δ βλέπουμε ε, τις χώρες αυτές υπό πρόγραμμα, πρόγραμμα το οποίο κατάρτισε η Τρόικα και έγινε αποδεκτό από τις χώρες. Τώρα, τα κριτήρια μπορούν να ήταν διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μας ε, ε, ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο ήταν εθελούσια η συμμετοχή ή όχι αλλά εν πάση περιπτώσει ε, όλοι συμφώνησαν, τα συμβαλόμενα μέρη δηλαδή, η Τρόικα και τα κράτη-μέλη. Σε σχέση με αυτή τη δυναμική κατανομής, δηλαδή το θέμα των προγραμμάτων διάσωσης και της ε, κρίσης, υπάρχει μια αιτιώδη συνάφεια και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς έχει αυτή η κατανομή. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό στον τομέα της απασχόλησης με πολλές ε, διαρθρωτικές παλινοδίες στον κοινωνικό τομέα με συνέπειες κατά των νέων όπου μπορούν να ανακύψουν και συγκυριακά προβλήματα πέρα από τα οικονομικά. Και που οδήγησαν σε πολλές ε, παλινοδίες κατά των νέων και διαφυγή εγκεφάλων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα 25% των ε, νέων έχει αποχωρήσει από τις χώρες όπως είδαμε στην περίπτωση της Ιρλανδίας. Και Ακόμα και αν υπάρχουν ρυθμοί ανάπτυξης, χρειαζόμαστε μία δεκαετία για να φτάσουμε σε επίπεδα απασχόλησης που είχαμε πριν από τα προγράμματα διάσωσης. Άρα, συμπεράναμε όλοι ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό, έχουν έχει πληγεί ο πληθυσμός, έγιναν σφάλματα με καλή καλή την πίστη βεβαίως, παρά την καλή θέληση, όμως έχουν γίνει λάθη. Δεν είχαμε σωστές μελέτες, αυτό σχεδιάσαμε και επειδή δεν εισακούστηκαν άνθρωποι που θα έπρεπε σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικών ζητημάτων. Στις ακροάσεις δεν ζητήσαμε την άποψη του ΔΟΕ, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Επιτροπής Απασχόλησης, της ΕΟΚΕ. Δεν έγινε διαβούλευση με κανέναν η Τρόικα έλαβε αποφάσεις χωρίς ε, προγενέστερες μελέτες για να καταπραίνουν τις συνέπειες. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν ο τραπεζικός τομέας, αλλά δεν σεβαστήκαμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Επίσης μπήκε στη γωνία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να έχουμε επηρεάσει για να διορθωθούν τα σφάλματα, όμως βρισκόμασταν σε κατάσταση οστρακισμού. Η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη βεβαίως και δεν απέτυχε, αλλά δυστυχώς έγιναν πολλοί αυτοσχεδιασμοί. Μιλήσαμε για χρονοδιαγράμματα ανάκτησης δυνάμεων που οδήγησαν σε ευθύνουσα πορεία της ανάπτυξης και το θέμα των διαρθρωτικών ελλημάτων δεν λήφθη υπόψη σοβαρά. Άρα καταστράφηκε ο κοινωνικός ιστός και ο κοινωνικός διάλογος διαγράφει. Οι συστάσεις είναι σημαντικές. Εγώ δεν καταφέρομαι κατά κανενός, αλλά με βάση τα σφάλματα που έχουν διαπραχθεί, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ανακτήσουμε δυνάμεις έτσι ώστε οι κοινωνικές συνέπειες να μην είναι τόσο δραματικές όσο είναι μέχρι τώρα. Βλέπετε στους συμβιβασμούς από το α μέχρι το gg, ε, βλέπετε τις συστάσεις και ζητάμε το εξής, να γίνει μία μελέτη αντικτύπου. Έχετε την ε, ΕΟΚΕ την, το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, τον ΩΣΑ, ας ε, διενεργηθεί μία μελέτη για να δούμε τι συνέβη. Ποιοι επλήγησαν οι εργαζόμενοι, οι νέοι με τα προγράμματα αυτά διάσωσης για να γίνει μια σωστή διάγνωση. Ζητάμε λοιπόν από από την Επιτροπή να βοηθήσει αυτούς που ζουν μία δυσίωνη κατάσταση να μπορέσουν να ανακτήσουν δυνάμεις, ιδιαίτερα οι νέοι, έτσι ώστε να προωθήσουμε τον κοινωνικό διάλογο που έχει καταστραφεί στις τέσσερις αυτές χώρες. Και θα πρέπει να διορθωθούν τα ε, ε, σφάλματα και όχι να τα δεχτούμε ό,τι και να έγινε. Τα προγράμματα πρέπει να λήξουν το συντομότερο δυνατόν. Έληξε το πρόγραμμα της Ιρλανδίας, αλλά θα πρέπει να ισχύσει και για τις άλλες χώρες με εναλλακτικά δηλαδή προγράμματα. Να είναι ευρωπαϊκά προγράμματα όπου να σχετίζονται, να συμμετέχουν όλα τα θεσμικά όργανα και όχι να μας λένε οι εξωευρωπαϊκοί παράγοντες πώς να διασωθούμε. Να είναι προγράμματα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση όπου να ακούμε τους κοινωνικούς εταίρους και να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις επιπτώσεις και να σεβόμαστε τις ε, ε, διεθνείς ε, συμφωνίες αυτό αφορά και το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, τον ΩΣΑ και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να πλήξουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα ούτε τις διεθνείς μας συμφωνίες. Τέλος, Πρόεδρε, ζητούμε μία για πάντα να εξισορροπηθούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές κατά συνετό τρόπο εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού ε, στόχου. Αυτό αφορά το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ βέβαια. Και επίσης δεν θα βγούμε από αυτή την κρίση αν δεν δημιουργηθεί απασχόληση. Αν δεν υπάρξουν έσοδα δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Θα πρέπει να ανακτήσουν δυνάμεις οι ΜΜΕ, να προωθηθούν οι πιστώσεις και ε, να προωθηθεί η προσφορά για να υπάρχει και ζήτηση. Να προωθήσουμε προενεργές πολιτικές απασχόλησης και να βοηθήσουμε τις πιο ευάλωτες ομάδες. Ε, να εγγυηθούμε την απασχόληση για τους νέους, γιατί αν χάσουμε αυτή τη γενιά θα υπάρχουν ολέθριες συνέπειες, αλλά θα έχουμε χάσει και κάθε διάλογο με το μέλλον. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαρκάς, τον εισηγητή για τις επιπτώσεις του έργου της Τρόικας. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Αρχικά έχουμε την κυρία Ρεγίνα Μπάστος, σκιώδης από πλευράς του ΕΛ και μετά Μαριάννη Ναρκίν για την ΑΛΔΕ. Κυρία Μπάστος, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πολύ για όσα προείπε ο κύριος ε, Θέρκας, για τα φιλικά του λόγια τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Είχαμε μία δύσκολη συνεργασία γιατί το αρχικό σχέδιο ε, είχε, ενείχε ιδιαίτερα δραματικά στοιχεία και επιθετικούς ε, προσδιορισμούς. Εμείς θεωρήσαμε ότι πρέπει να είμαστε προπάντων επικοδομητικοί, γι' αυτό στην αρχή η οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες, αλλά μετά με την συνάντηση των σκιωδών ε, βρήκαμε μία γέφυρα συνεργασίας εκμεταλλευτήκαμε τα αρχικά στοιχεία και αποβάλαμε τα, εκμεταλλευτήκαμε τα θετικά στοιχεία και αποβάλαμε τα τοξικά. Ε, έτσι ώστε να υπάρχει μια επικοδομητική θεώρηση. Φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και έτσι φτάσαμε σε κείμενα σε 32 συμβιβασμούς που υποστηρίζει το ΕΛΚ και ο τελικός στόχος ο τελικός στόχος είναι ρεαλιστικός και αντικειμενικός. Όπως ήδη προελέχθη, προσπαθήσαμε να μην είμαστε επιθετικοί, ιδιαίτερα επιθετικοί κατά της Τρόικας, δηλαδή να μην την στήσουμε στον τοίχο, αλλά να προωθήσουμε μία ε, ρεαλιστική θεώρηση με μηνύματα και διδάγματα για το μέλλον με βάση την εφαρμογή του σύμφωνου αυτού χρηματοοικονομικής βοήθειας για τις τέσσερις αυτές χώρες. Ο βασι... Η βασική σχετίζονται με την κατάσταση των τεσσάρων χωρών πριν από την έλευση της ε, Τρόικας και μετά με τα προγράμματα ε, διάσωσης για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία αυτό των ε, τεσσάρων χωρών. Οι τέσσερις χώρες ε, ζήτησαν προγράμματα διάσωσης, ζήτησαν τη βοήθεια αυτή και δεν επευλήθησαν τα προγράμματα αυτά από την Τρόικα. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι τα κράτη δεν είχαν άλλες εναλλακτικέ από το να δεχτούν την μονομερή ε, επέμβαση, η παρέμβαση της Επιτροπής της ΕΚΤ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή οι χώρες αυτές ε, βρίσκονταν σε ολέθρια κατάσταση και χρειάστηκε να ζητήσουν χρηματοοικονομική βοήθεια. Μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος έτσι ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τη λειτουργία της κρατικής μηχανής και της δημόσιας διοίκησης, του συστήματος υγείας, της εκπαίδευσης, της καταβολής συντάξεων και μισθών, γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν. Επίσης υποστηρίξαμε ότι όταν παρενέβη η Τρόικα, οι χώρες αυτές ε, ήταν ιδιαίτερα ευάλωτες και εάν δεν εφαρμόζονταν αυτά τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής, η κατάσταση θα ήταν ακόμα πιο ολέθρια, ιδιαίτερα σε κοινωνικό επίπεδο. Επίσης, δεν αρνούμαστε τα αυταπόδεικτα στοιχεία που τόνισε ο εισηγητής, ότι δηλαδή σε επίπεδο απασχόλησης οι συνέπειες ήταν καταστροφικές, ιδιαίτερα ως προς την ανεργία των νέων και είχαμε και την πίεση χρόνου παράλληλα. Είχαμε απειροελάχιστο χρόνο για να αντιδράσουμε και να εφαρμόσουμε αυτά τα προγράμματα ε, βοήθειας και διάσωσης. Δεν αρνούμαστε όμως ότι αυτές οι αρνητικές συνέπειες που αισθάνθηκαν τα κράτη-μέλη ε, δίνουν δειλές θετικές ενδείξεις, δηλαδή αύξηση της απασχόλησης, μείωση της ολικής ανεργίας, ε, θετική έκβαση των διαρθρωτικών ε, μεταρρυθμίσεων και επίσης σε αντίθεση εκτός και απορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στη δική μου χώρα, στην Πορτογαλία, λάβαμε υπόψη τις ευάλωτες κατηγορίες, ε, ιδιαίτερα τους μικροσυνταξιούχους, του και τους ανέργους έτσι ώστε να, έχουν, να λάβουν ειδικά επιδόματα. Επίσης, ο κοινωνικός διάλογος δεν προωθήθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη αντίθετα. Ορισμένα κράτη κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τα κύρια συνδικάτα για να φτάσουν σε κοινωνική ειρήνη η οποία επιβάλλεται κατά την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων κοινωνικής προσαρμογής. Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα θεσμικά όργανα είχαν να αντιμετωπίσουν μια κρίση χωρίς προηγούμενο δηλαδή με δυνατότητες ε, δράσης ε, πολύ περιορισμένες βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα χωρίς να μπορέσουν να αντιδράσουν και έπρεπε να εξεύρουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Και τα θεσμικά όργανα δεν ήταν έτοιμα. Παρόλα αυτά προσπαθήσαμε να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες και δεν υπήρχε και καμία νομική βάση που να επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή είχαμε να κάνουμε με απρόβλεπτες καταστάσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε στην επόμενη αυτή διαδικασία θυσιών των πολιτών μας, που οι πολίτες υπέστη καν υπέστησαν, με συγχωρείτε, ε, στοικά. Άρα η έκθεση αυτή είναι εξισορροπημένη, πολύ αντικειμενική, χωρίς ε, να είναι ε, ιδεολογικά φορτισμένη. Γι' αυτό και το ΕΛΚ με μεγάλη χαρά θα υπερψηφίσει αυτή την έκθεση διότι είναι καρπός ε, μίας ε, διεργασίας και συνεργασίας των δύο μεγάλων ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μπόστος. Το λόγο έχει η Μαρία Αρκίν, σχεώδης από πλευράς ε, της Άλντε. Κυρία Χάρκιν, ευχαριστώ πολύ. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του, αλλά και για την ε, διάθεση που επέδειξε, την οποία θεωρώ πραγματικά εξαιρετική. Τη βούλησή του ε, να εξευρεθεί ισορροπία, συμφωνία και συμβαστικές λύσεις. Νομίζω ότι ήταν ε, εξαιρετικά χρήσιμη και επικοδομητική στάση του και τον ευχαριστώ. Είχαμε κάποιες ε, περαιτέρω επαφές και σήμερα. Υπάρχουν ακόμα κάποια ζητήματα με κάποιους από τους συμβιβασμούς. Έχουμε πέσει βέβαια σε λίγα μόνο σημεία. Έχουν μειωθεί τα σημεία προβληματισμού και έχω και κάποιες γενικές παρατηρήσεις για την ίδια την έκθεση. Μας ε, προβληματίζει ε, ο συμβιβασμό FF στο πεδίο 5, όπου μία από τις συστάσεις που μας δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί όταν μιλάμε για συλλογικέ συμβάσεις, τις οποίες και εμείς βεβαίως στηρίζουμε, τότε δεν θέτουμε ε, προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Μιλάμε για συλλογικέ συμβάσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι έτσι τίθεται ένα πρότυπο που η Άλντε εν γέννη δεν μπορεί να στηρίξει. Από εκεί και πέρα μας δημιουργεί πρόβλημα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης. Υπάρχουν εθνικές βεβαίως τέτοιες υπηρεσίες, όμως το θέμα είναι ότι δεν έχουμε αφήσει τις συλλογικέ συμβάσεις μόνο, ε, έχουν τεθεί ως προαπαιτούμενο το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το πραγματικό νόημα των συλλογικών συμβάσεων. Μετά, για την ε, συμβαστική CC αναφέρεται ότι καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντα υπόψη τις θυσίες ε, που έκαναν αυτές οι χώρες, να παράσχουν ε, στήριξη μετά την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων και μέσω επαρκών χρηματοδοτικών ε, μέσων για την κάλυψη των αναγκών τους και ούτω Θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Ο εισηγητής πώς ακριβώς θεωρεί θα καλυφθούν αυτές, ε, αυτοί οι επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι, από πού θα προκύψουν, εφόσον μόλις έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν υπάρχουν ε, και πολλά κοινωνικά κονδύλια, τα περισσότερα μάλιστα έχουν ε, ήδη διατεθεί, ή μάλλον έχει αποφασιστεί πού θα διατεθούν, επομένω δεν μένουν ακόμα πολλά αδιάθετα. έχει υπάρξει διατύπωση της συμβαστικής ζήτα, περιμένουμε να τη δούμε. Και τέλος για την ΕΕ, ζητήσαμε από τον εισηγητή στο τελευταίο τμήμα του ΕΕ να έχουμε την ίδια διατύπωση που είχαμε στο AGS. Και αυτό σίγουρα θα μας βοηθήσει να στηρίξουμε. Ξέρω ότι κάποια μέλη μας έχουν πρόβλημα με το πρώτο τμήμα του κειμένου, εγώ προσωπικά δεν έχω. Όμως ε, θα θέλαμε πραγματικά να αναφέρονται τα όσα αναφέρονται στην ε, ετήσια έκθεση προόδου. Όμως πραγματικά θα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την επικοινωνική του στάση, το πνεύμα συμβιβασμού, Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων. Μια άλλη παρατήρηση που θα θέλω να κάνω σύντομα είναι ότι αυτή η έκθεση αφορά ε, τον ρόλο και τη λειτουργία της ε, Τρόικα. Δεν μιλάμε για το τι συνέβη προηγουμένως, μιλάμε για τα αποτελέσματά της. Υπήρξαν ε, βεβαίως διαφορετικές καταστάσεις στα επιμέρους κρατημέλη και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ενώ τα κράτη-μέλη ζήτησαν τη συνδρομή αυτών των θεσμικών οργάνων, εδώ μιλάμε για μη εθελοντική ε, μετανάστευση για παράδειγμα και για κάποια κράτη-μέλη σας διαβεβαιώ ότι ε, παρά τη θέλησή τους ζήτησαν την ε, συνδρομή αυτών. Εμείς δεν είχαμε άλλη επιλογή, έπρεπε να σώσουμε το τραπεζικό σύστημα, έπρεπε να δώσουμε 64 δις για να σωθούν οι τράπεζες, αλλιώς θα είχε μεταδοθεί η, η κατάρρευση αυτή και σε άλλες χώρες θα, είχε, θα είχαμε οδηγηθεί σε ολοκληρωτική καταστροφή και κατάρρευση και γι' αυτό μας ε, βοήθησε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μας δάνεισαν αυτά τα χρήματα με επιτόκιο 6% γιατί ε, ανακεφαλοποιήσαμε τις τράπεζες και κοινωνικοποιήσαμε το χρέος. Όταν να πούμε δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη εθελοντικά ε, με την ίδια βούληση ζήτησαν αυτή την αρρωγή είναι λίγο τραβηγμένο. Όμως, ε, να είμαστε δίκαιοι, στην Ιρλανδία έγιναν προσπάθειες ε, να μην αυξηθούν οι ανισότητες ε, στο κοινωνικό μας σύστημα. Όμως οι πρόσφατες εκθέσεις του ΩΣΑ δυστυχώς δείχνουν ότι περισσότερο επλήγησαν οι πλέον πλουσιότεροι και οι πλέον φτωχότεροι των κοινωνικών στρωμάτων. Βεβαίω, οι πιο πλούσιοι είναι αυτοί που μπορούν να επιβιώσουν ενώ οι φτωχότεροι όχι τόσο εύκολα. Συμφωνώ με τη Ρετζίνα Βάστος ότι σίγουρα βρεθήκαμε στο μάτι του κυκλώνα χωρίς άλλη λύση. Όμως αυτό σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, αλλά σε σημαντικό βαθμό, ο λόγος ήταν ότι ε, ήμασταν τμήμα μιας ευρωζώνης ε, που δεν μας τέριαζε και οι πολίτες ε, ζημιώθηκαν περισσότερο από αυτή την κατάσταση. Τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι αυτό το θέμα δεν έχει λυθεί ακόμα. Ξέρω ότι είναι προ το οικονομικό ζήτημα, όχι ζήτημα απασχόληση, αλλά βρισκόμαστε ακόμα μέσα αυτό το νόμισμα, την νομισματική ένωση, με τεράστια πλεονάσματα σε κάποιε χώρε, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν τεράστια λύματα αλλού. Νομίζω ότι δεν, έχουμε, δεν είμαστε ακριβώ στο μάτι του κυκλώνα, όμω δεν έχουμε προχωρήσει και πολύ δεν έχουμε διαφύγει εντελώ το κίνδυνο. Και πάλι ευχαριστώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Χάρκινγκ. Μαρία Κορνέισεν από πλευρά των ε, οικολόγων Πρασίνων, ο Σοσκιώδης και μετά ε, Εντίθε Στρέλια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Σε κάποιες ε, συναντήσεις των σκιωδών παρευρεθήκαμε κι εμείς που δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολες, όμως τελικά καταλήξαμε σε συμβαστικέ τροπολογίε με τι οποίε οι περισσότεροι μπορούμε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε. Θέλω και εγώ να συμφωνήσω με τη Μάριαν Χάρκιν. Σε πολλά από όσα είπε, τουλάχιστον στα τελευταία δύο-τρία σχόλιά τη, ε, για την ε, μη εθελοντική συμμετοχή των κρατών μελών σε αυτά τα προγράμματα ελπίζω πραγματικά αυτό τουλάχιστον να ενσωματωθεί στην Επιτροπή της ΕΚΟΝ, γιατί πολλά πήγαν στραβά. Και βεβαίως θα πρέπει ε, να ε, πούμε ποιος φέρει ευθύνη, αλλά θα πρέπει να καταδείξουμε και τους πραγματικούς υπέτειους το δύσκολο σε αυτές τις ε, συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών ήταν να, να γίνει μια εξισορρόπηση, να ε, αναφέρουμε τα ονόματα αυτών των χωρών, αλλά να διατηρούμε και μια ισορροπία. Και τελικά είπαμε κάποιες χώρες, ορισμένες χώρες, οι περισσότερες χώρες σε πολλές παραγράφους. Εγώ θα προτιμούσα να κατανομάσουμε αυτές τις χώρες. Αλλά και αυτό είναι δύσκολο. Γιατί ενώ στην Πορτογαλία υπάρχουν πράγματι μικρότερες ε, κοινωνικές ανισότητες και μικρότερο κίνδυνος ε, φτώχειας από ότι τα υπολοιπα κρατημέλη, είναι δύσκολο αυτό να το ε, θέσουμε σε στοιχεία, γιατί δεν έχουμε και πολλά αξιόπιστα στοιχεία για αυτή την κατάσταση ή τουλάχιστον έρχονται καθυστερημένα. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε αφορούν την κατάσταση πριν από δύο χρόνια. Είναι λοιπόν δύσκολο νομίζω ότι θα πρέπει να ε, καταρτήσουμε μία έκθεση που να είναι επικριτική απέναντι στην ε, Τρόικα. Θα έπρεπε να επικεντρωθούν περισσότερο και στην ε, κοινωνική ε, πτυχή. Να έχουμε δηλαδή κατά νου ότι αυτά τα χρήματα, τα επιδόματα, οι συντάξει που κόβονται είναι τα χρήματα που χρειάζεται ο κόσμος για να ζήσει. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρξει ευρία πλειοψηφία για την έκθεση. Εξίσου σημαντικό όμως είναι να ε, διαβιβαστεί ένα ισχυρό ή τουλάχιστον ένα μήνυμα. Από ό,τι φαίνεται προς το παρόν, η ε, αντίστοιχη έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την Τρόικα είναι πολύ πιο επικριτική από τη δική μας και εστιάζει περισσότερο την προσοχή της ε, στις επιπτώσεις της δράσης της Τρόικας. Πρέπει και εμεί λοιπόν να κοιτάξουμε τι κάνουν εκείνοι και να φροντίσουμε να κοιμαρθούμε και εμεί στο ίδιο μικρο κύματο. Όχι να είμαστε τόσο λιγότερο επικριτικοί από εκείνοι. Θα ήθελα σε αυτό το πνεύμα να υπερψηφίσουν τις τροπολογίες 2.14 ε, και 2.35 οι υπόλοιπε πολιτικές ομάδες. Και τελευταία παρατήρηση για την ισορροπία που χρειάζεται να έχουμε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες που έχουν πλεονάσματα θα πρέπει να ε, κάνουν κάποιες προσπάθειες να μειώσουν τα πλεονάσματα και να εξευρεθεί νέα ισορροπία. Και γι' αυτό έχουμε επισημάνει, αυτό έχουμε επισημάνει και στην τροπολογία 240 που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κορνέλισεν. κυρία Στρέλια για το λόγο. Και κλείνει εδώ ο κατάλογος Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα συνενετικό πλαίσιο λειτουργίας, κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο. Είναι εξισορροπημένη η έκθεση και ε, ρεαλιστική. Αυτά προελέχθησαν σε σχέση με την εργασία του εισηγητή. Αλλά μία ρεαλιστική έκθεση θα πρέπει να ε, ερμηνεύσει αυτή την τραγική κατάσταση που ζουν οι πολίτες. Πολλοί έχασαν την επιχείρησή τους, άλλοι το σπίτι τους, άλλοι το εργοστάσιό τους, άλλοι την εργασία τους και άλλοι έχασαν και τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Είδα να, να συρρυκνούνται τα έσοδά τους. Είχαμε μία κοινωνική ε, επιδίνωση ε, στις χώρες αυτές υποδιάσωση. Κάτι το οποίο αναγνώρισε και η ίδια η Τρόικα η οποία αναγνώρισε ότι υπήρξαν πολλά σφάλματα στη συνταγή αυτή της ε, λιτότητας και φτάσαμε σε πολλά άκρα ε, παρά τις συστάσεις ε, πολλών οικονομολόγων που είχαν λάβει ακόμα και το βραβείο Νόμπελ. Εν πάση περιπτώσει είχαμε να κάνουμε με εθνικές επιλογές και πολλές φορές ε, δεν υπήρχαν και περιθώρια στη δική μου χώρα, στην Πορτογαλία. Έχουμε μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, με αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και έλλειψη επενδύσεων σε τομείς όπως η έρευνα, υγεία, εκπαίδευση. Καθίσταται σαφές ότι οι κοινωνικές επιπτώσεις της ε, παρέμβασης της Τρόικας θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να οδηγήσουν σε επιθυμητά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, σε μία χώρα 10 εκατομμυρίων το 2012 μετανάστευσαν 120.000 Πορτογάλοι γιατί δεν είχαν απασχόληση. Άρα τώρα να λέμε ότι ο δείκτης απασχόλησης ίσως έχει μία ελάχιστη ανωδική τάση δεν σημαίνει τίποτα. Διότι δεν μειώθηκε πραγματικά μειώθηκε ο ενερικός ε, πληθυσμός, διότι πολλοί αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν και αποθαρρύνθηκαν. Εκείνοι που είχαν χάσει κάθε ελπίδα να μπουν στην αγορά εργασίας. Στους νέους η κατάσταση είναι πολύ επώδυνη. Έχουμε έναν υψηλότατο δίκτυ ανεργίας. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για να πιστεύουν οι άνθρωποι σε μας, διότι έχουμε ευθύνη έναντι των εκλογέων μας και δεν θα πρέπει να χρυσώσουμε το χάπι ε, και να μην αναγνωρίσουμε τον ολέθριο ρόλο της Τρόικας. Πολλοί νέοι έχασαν την εργασία τους ή δεν τη βρήκαν καν και γι' αυτό θα πρέπει πρωτίστως να δώσουμε ελπίδα στους νέους για να πιστέψουν στην Ευρώπη και τα θεσμικά μας όργανα. Αυτό είναι η πρώτη στη υποχρέωσή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξαναδίνω το λόγο στον εισηγητή, στον Αλεχάνδρο Θέρκας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα τα σχόλια, τα θετικά και τα λιγότερα θετικά, λιγότερο θετικά. Αναγνωρίζω τις επικρίσεις. γιατί ήθελα να συνεργαστώ με όλους. Πολλά δεν μπορούσαν να τα δεχτούν η Ρετζίνα ή η Μαρία Χάρκιν. Οι συμβιβασμοί αυτοί αποτελούν τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Γι' αυτό φτάσαμε και σε αυτή τη συμφωνία. Ε, αύριο θα δούμε κατά πόσο και πολλές άλλες τροπολογίες των ομάδων θα περάσουν. Εγώ θα υποστηρίξω τις ε, τρεις ε, τροπολογίες των πρασίνων. Θα υποστηρίξω και τις τρεις. Για να απαντήσω στη Ρετζίνα, δεν ήθελα να μπω σε μια ιδεολογική συζήτηση, αλλά σε μια ρεαλιστική και επικοδομητική παρά τις διαφορετικές θέσεις που έχουν οι δύο βουλευτές από την Πορτογαλία. Θα μπορούσε να γίνει μια ελληνική συζήτηση, μια ιρλανδική, μια πορτογαλική και μια ισπανική. Θα πρέπει να δούμε τα κοινά στοιχεία όμως και να βρούμε κοινέ λύσεις. Πολλές φορές έπρεπε να δώσουμε παραδείγματα αλλά δεν κάναμε μία ανάλυση χώρα προς χώρα. Βρίσκουμε τα κοινά στοιχεία που διέπουν και τις τέσσερις χώρες. Εγώ αναγνωρίζω την μείωση της απασχόλησης κατά 15% σε όλες τις χώρες. Αυτό είναι, αυτό είναι το ελάχιστο αλλά βλέπουμε μία απειροελάχιστη ανωδική πορεία του δίκτυ. Μιλάμε για ελάχιστα δεκαδικά. Ε, ήρθαμε και σε επαφή με τη ε, Eurostat. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερος ο χρόνος, αλλά θέλησα να καθησυχάσω την Edith Estrella. Γιατί δεν πρέπει να συγχέουμε την ανεργία με τις θέσεις εργασίας πάντα. Ξέρουμε ότι γίνεται μαζική έξοδος των εργαζόμενων, κάτι το οποίο στρεβλώνει τα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή βελτιώνει τους δείχτες, αλλά ο ενεργός ε, πληθυσμός ε, είναι ε, λιγότερος. Αλλά στην περίπτωση της Πορτογαλίας της Ελλάδας και της Κύπρου βλέπουμε μία απειροελάχιστη ανωδική πορεία του δίκτυ απασχόλησης. Γι' αυτό δεν ήταν ιδεολογική συζήτηση, ήταν συζήτηση ουσίας. Σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Χάρκιν, ε, δέχομαι τη συνετή της θέση ξέρω πώς επλήγει η χώρα της. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το δημόσιο χρέος ήταν τραπεζικό χρέος, το οποίο ανέλαβε ο Ιρλανδικός λαός. Άρα αναγνωρίζω ότι η κατάσταση ήταν πολύ σκληρή. Ως προς τις τροπολογίες της, έχουμε έρθει σε συμφωνία με τους ε, φιλελευθέρους, αλλά όχι σε όλα τα στοιχεία. Στο FF μιλάμε για το ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ενδεχόμενη αύξηση των μισθών. Διότι κυρία Χάρκιν όλοι έχουμε πληγή σε σχέση με, το θέμα ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το νόμισμά μας, γιατί έχουμε κοινό νόμισμα. Επειδή όμως υπάρχει αποπληθωρισμός και μείωση των ε, μισθών, υπήρξαν ολέφριες συνέπειες και στις επιχειρήσεις θα δούμε ποια θα είναι και η τάση των εξαγωγών, αλλά το 80% εξαρτάται από την εσωτερική ζήτηση, η οποία έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό θα πρέπει να μην ακολουθήσουμε αυτή την ατραπό της ε, μείωσης ε, της εσωτερικής ζήτησης. Αν δεν αυξηθούν μισθοί, δεν θα υπάρχει και εσωτερική ζήτηση. Άρα θα πρέπει να αλλάξει ο προσανατολισμός μας για το μέλλον. Γι' αυτό δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το τμήμα του FF. Τώρα για την ανάκτηση της δημόσιας υγείας, εκπαίδευσης, την αντιμετώπιση της φτώχειας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Επιτροπή και το ΕΚΟΦΗΜ βρήκανε 500 δις για να σώσουν τις τράπεζες, δεν μπορούν να κάνουν κάτι για να σωθούν τα παιδιά και οι φτωχοί. Θα μπορούσα να ε, δεχτώ τη λέξη sufficient, επαρκής, που είναι στην πρότασή σας, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν χάσει κάθε ελπίδα. Δηλαδή να χτυπήσουμε την φτώχεια των ανηλίκων και να βοηθήσουμε την υγεία, την εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Πρόκειται για ένα ε, καθόλου ε, ανυπέρβλητο ζήτημα αν, λάβουμε υπόψη και αν σκεφτούμε την τραπεζική κρίση και πώς αντιμετωπίστηκε, θεωρώ ότι θα πρέπει να βρεθούν ε, πόροι για να αντιμετωπιστεί η κοινωνική κρίση. Τώρα, η τροπολογία ε-ε εμένα μου αντιμετωπίζει, μου δημιουργεί, με συγχωρείτε, ένα πρόβλημα. Το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ θα πρέπει να συμφωνήσει με το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Αυτό δεν αρέσει στον Όλυ Ρεν. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο Συμβουλίων ε, ΕΠΣΚΟ και ΕΚΟΦΗΝ. Δεν λέω ότι η δική μας έκθεση έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη σημασία από την έκθεση της ΕΚΟΝ. Η Ρεζίνα Μπάστος ε, συμμετέχει και στις δύο επιτροπές. Εμείς προσπαθούμε να δείξουμε κατανόηση, αλλά δεν φτάσαμε ποτέ στα άκρα. Εγώ είμαι ακόμα και πιο, μετριοπαθής και από τον κύριο Κάρας. Θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Βρίσκομαι στο τέλος της πολιτικής, της πολιτικής μου σταδιοδρομίας. Εάν δεν μειωθεί το χάσμα που υπάρξει μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων, τότε θα αποτύχουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδρασε σαν να ήταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, σαν να ήταν τραπεζίτες. Δεν πρέπει να το κάνουμε και στο μέλλον, να γίνουν τα ίδια ε, ε, σφάλμα. Η γλυκιά λοιπόν, η γλυκύτατη ε, ρεζίνα μπάστος θα πρέπει να μην είναι τόσο σκληρή απέναντί μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήγητη. Τα σημειώνουμε όλα αυτά. Θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί στην Επιτροπή Απασχόλησης και η έκθεση θα περάσει στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Προτείνω τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο, υπάρχει μόνο 8. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τις απαλλαγές. Θα ξεκινήσουμε με τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και θα γίνει κοινή συζήτηση για το σύνολο των ε, απαλλαγών. Γενικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έκθεση σχετικά με την απαλλαγή σε όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού των οργανισμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό έτος 2012, επιδόσεις δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος, σημείο μετά 10 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη τη Επαγγελματική Κατάρτιση, ΕΝΤΕΦΟΠ. 11. Απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεω και Εργασία. Σημείο 12. Απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ιδρύμα Επαγγελματική Εκπαίδευση. Και σημείο 13. Απαλλαγή 2012 για το Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το σύνολο αυτών των απαλλαγών. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μπερέ, που δεν βρίσκεται εδώ σήμερα. Και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Θέρκας, ο οποίος την αντικαθιστά. Θα ήθελα να είμαι σύντομος, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να σας διαβάσω εντάχει τη δήλωσή της. Καταρχήν ε, θα ήθελα να ζητήσει συγγνώμη, σήμερα δεν μπορούσε να παρευρεθεί και θα ήθελε να ευχαριστήσει τους πάντες που την βοήθησαν για τη διαδικασία απαλλαγής αυτών των οργανισμών. Θεωρεί ότι αύριο θα εγκριθούν και θα προβάλλει τρεις τροπολογίες συμβιβασμού. Θα ήθελε στο τμήμα 3 της Επιτροπής να προβάλλει μία τροπολογία συμβιβασμού ε, με βάση μία ιδέα του Τσάμπα Όρη για να ε, προσβλέπουμε σε απλουστευμένες, απλοποιημένες διαδικασίες στο μέλλον. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Επίσης θα ήθελε να ψηφιστεί ένας συνδυασμός για τις τροπολογίες 2, 3 και 4 των Τσάμπα Όρη και Μαρία Χάρκιν όπου ε, αναγνωρίζουμε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών, όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια με τα πρωτόκολλα, τα σχέδια εκπαίδε... Ε, ε, έρευνας, με συγχωρείτε, σε σχέση με τους τέσσερις, τέσσερις οργανισμούς και ιδρύματα, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Και τέλος, η κυρία Μπέρες θα ήθελε, σε σχέση με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, να λάβει υπόψη τα σχόλια του ελεγκτικού συνεδρίου για ένα πρόβλημα που ανέκυψε. Δηλαδή, οι λειτουργικές ε, πιστώσεις είναι πολύ υψηλές μέσα στα πλαίσια της έγκρισης του προϋπολογισμού. Αλλά ίσως να είναι τεχνική υφή στο θέμα και δεν θα ήθελε να αμφισβητήσει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Θα ήθελε ο κύριος Τσάμπα Όρη στην πρώτη παράγραφο να αλλάξει το κείμενο. Το το request να ε, αλλάξει με το ask. Αντί requests, asks. Για να φαίνεται ότι πρόκειται για μία διασάφηση και για να μην, αλλάξει το, να μην αλλάξουν οι σχέσεις μας με το επαγγελματικό αυτό κέντρο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σέρκας. Ο κύριος Ερή, σκιώδης συζητητής πολευράς του ΕΛΚ, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε. Τελευταία φορά νομίζω συζητήσαμε όλα τα σημαντικά θέματα, επομένω θα είμαι σύντομος. Σε ό,τι φορά την τροπολογία που κατέθεσα, από ό,τι φαίνεται ένα τμήμα της τροπολογίας γίνεται αποδεκτό, παραμένουν κάποιες ε, διαφορές απόψεων. Θα δούμε τι θα γίνει στην ψηφοφορία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη ΣΕΝΤΕΦΟΠ, μιλήσαμε για αυτή την τροπολογία, ανταλλάξαμε διάφορα email. Αν θέλετε μπορούμε να καταστήσουμε το request με το ask. Αν θέλετε να βάλουμε ask στο κείμενο, να ρωτήσουμε, να ζητήσουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, μπορούμε να αποδεχθούμε από αυτή την πρόταση και έτσι μπορούμε να περάσουμε με, αυτή την, με αυτό το συμβασμό στην ψηφοφορία. Ωραία, να επαναλάβω για τον κύριο Σέρκας. Α, εντάξει. Δέχεται ο σκιώδης συζητητής να αλλάξει το request και να γίνει ask. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ρή. Η κυρία Χάκινγκ το λόγο σκιώδης εισηγήτρια από πλευράς Άλντε. Ευχαριστώ. Ε, όπως και ο κύριος Ερή μπορώ να είμαι και εγώ πολύ σύντομη διότι συζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση τα βασικά θέματα και συμφωνήσαμε στους συμβιβασμούς και δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ. Merci Ευχαριστούμε την κυρία Χάρκιν. Δεν ζητά κανείς άλλο στο λόγο. Ο κύριος Σέρκας σημείωσε τη Συμφωνία των Φιλελευθέρων και του ΕΛΚΑ για αυτό το αίτημα. Επομένω, ε, κλείνει και αυτό το ζήτημα. Ε, ε. Ψηφοφορία θα γίνει αύριο στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού θα γίνει στις 17 Μαρτίου και στην Ολομέλεια στη Σύνοδο του Απριλίου. Ας κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Ah euh, euh, διακοπή ενός λεπτού λοιπόν για να δούμε αν η κυρία Στάκοβα θα φτάσει στην αίθουσα για να περάσουμε στο σημείο 14. για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην κοινότητα. So, dear colleagues, we can start again. Um, Ωραία, συνάδελφοι, ας ε, συνεχίσουμε τώρα. Σημείο 15 της ημέρης διάταξης, σε πρόταση οδηγίας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ναυτικούς που τροποποιεί τις οδηγίες 2008 2009, 2002 και 2001. Θα δώσουμε τώρα το λόγο απευθείας στην εισηγήτρια κυρία Ροντζούλη. The floor is yours. Grazie, grazie Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη για την αναμονή. Θα σας μιλήσω για τις τροπολογίες που ε, λάβαμε τις τελευταίες ε, ημέρες και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν υποβληθεί 18 τροπολογίες, πολλές εκ των οποίων δεν με βρίσκουν σύμφωνοι σε σχέση με το κείμενο που υπέβαλα, διότι το ανατρέπουν. Θεωρώ ότι το κείμενο αυτό είναι αρκετά συνεκτικό και ισορροπημένο όπου ε, ορίζουμε τις σωστές ε, κοινωνικές καλύψεις και ασφαλίσεις των ε, ναυτικών, αλλά δεν πρέπει να, να τρέψουμε αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα. Πρόκειται για μια πρόταση που αφορά μια σωστή κάλυψη των ε, ναυτικών καθώς ε, και την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Θα αρχίσω από τις ε, θετικές τροπολογίες, γιατί είναι και πολύ λίγες. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν αυτές τις ε, θετικές ε, προτάσεις που εισαγάγουν και νέα στοιχεία χωρίς να τροποποιήσουν πλήρως το περιεχόμενο 14, 16, 17 και 18 από τη συνάδελφο Μπαλντακίνο. Και αναφέρομαι στη Διεθνή Σύμβαση, την Ήλο που μπήκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο του 2013, αφού ε, υπέγραψαν 30 χώρες. Μιλάμε για τις ελάχιστες προδιαγραφές κάλυψης και ασφάλειας. Πρόκειται για τροπολογία 14. Οι 16 και 17 αφορούν τη σύμβαση ήλο, ενώ η 18 αφορά την βελτίωση των συνθήκων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό ορίζει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Σε σχέση, σε σχέση με τις αρνητικές τροπολογίες, 15, 19 και 22, 26, 27 και 29 της συναδέλφου και πάλι Μπαλντακίνου. Οι 15 και 27 δεν μπορούν να τύχουν της υποστήριξής μου διότι ε, αφορούν την παρέκταση της οδηγίας 2002 ε, κάθετος 14. Όπως σας είπα τη, ως προς την οδηγία 2001 23 αφορά την ακίνητη περιουσία, αλλά δεν μπορεί να ισχύσει στην περίπτωση των πλοίων ή των σκαφών διότι σχετίζονται με την ε, σημαία, με σημαία ευκαιρίας ενδεχομένως. Και σε αυτή την περίπτωση οι ναυτικοί ίσως υπάγονται σε ένα εργασιακό καθεστώς που είναι πολύ διαφορετικό. Και θα ήταν υποχρεωμένοι να μεταφερθούν αλλού από τον εργοδότη. Οι συλλογικές συμβάσεις διαφέρουν από σημαία σε σημαία. Η πρόταση τροπολογίας αφορά μείωση της προστασίας των Ευρωπαίων ναυτικών και δεν θα ίσχυε σε περίπτωση νιολόγησης κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οδηγεί σε αθέμητο ανταγωνισμό. Η τροπολογία 19 συμβαδίζει με την γενικότερη ανακοίνωση ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, αλλά ε, ξεφεύγει από το πλαίσιο της οδηγίας. Το διαδίκτυο σε όλα τα πλοία θα σήμαινε ε, υπερβολικό κόστος και δαπάνη. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μια ειδική νομοθεσία. Η 22 δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου που παραμένει. Γιατί θα έπρεπε να κατακαιρματιστεί αυτός ο διάλογος. Η 2002 κάθετος 14 που αφορά την πληροφόρηση και τη διαβούλευση, οι διαδικασίες αυτές δεν τηρούνται. Δεν μπορούμε να στρεβλώσουμε το αρχικό κείμενο γιατί η προσέγγιση της οδηγίας είναι πιο εξισορροπημένη, λαμβάνοντας υπόψη τις θαλάσσιες μεταφορές. Δηλαδή, τη διαφορά χρόνου, την ασφάλεια στο σκάφος και την απομάκρυνση από την ακτή. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η διαβούλευση αυτή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη μεταφορά. Η 26, η τροπολογία 26, όπως προβάλλεται, θα επέτρεπε στους εκπρόσωπους των εργαζομένων να μπλοκάρουν την μεταφορά ενός πλοίου έτσι ε, ώστε να πλήξουν και τις θαλάσσιες ε, μεταφορές. Η πρόταση αυτή δεν είναι και τόσο μακρόπνοη. Δεν δημιουργεί δηλαδή ανάπτυξη σε αυτό το τομέα. Εάν όμως θέλουμε να σταματήσουμε ε, το πλοίο, τη μεταφορά του, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι υπέρ των εργαζομένων πολλές ε, φορές τα πλοία μεταπολούνται από έναν εφοπλιστή σε έναν άλλον, αλλάζει, το νιολόγιο, αλλάζει και η σημαία. Και ήδη υπάρχουν ε, συλλογικές συμβάσεις για συλλογικές απολύσεις εργαζομένων. Οι συλλογικέ συμβάσει είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Η τροπολογία 29 είναι παρόμοια της κυρία Ρεντέρ. Αν δεν κάνω λάθο, κινείται πέραν από τα όρια που προβλέπει η Επιτροπή, διότι ζητά εξαιρέσεις από ε, ε, εξαιρέσεις, παρεκκλήσεις μάλλον, από τις ίδιες τις ρήτρε εξαίρεσης. Κάτι το οποίο ε, θα σήμαινε σε περίπτωση μεταφοράς διαφορετικές συνθήκες εργασίας. Άρα όχι επαρκή κάλυψη των ναυτικών ενώ εμείς θέλουμε να νομοθετήσουμε για το ακριβώς αντίθετο, να προστατεύουμε περισσότερο τους ναυτικούς. Οι 13, 21, 23 και 25 της κυρίας Στρέντερ, καταρχήν η 13 ε, αφαιρεί ένα μέρος του κειμένου και οι ΜΜΕ δεν υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 21 επίσης αφαιρεί ένα μέρος του κειμένου και αποκλεί τη δυνατότητα να αποκλειστούν αυτές οι δραστηριότητες από την Οδηγία 2008 σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας και 23 και 25 αλλάζουν ολόκληρο το αρχικό κείμενο και δημιουργούν αμφιβολίες τις οποίες δεν χρειαζόμαστε πέρα από αυτές που έχουμε. Οι 20, οι 24 και οι 20, 24 και 29 της κυρίας Μπερές. Η 20 δεν χρειάζεται, διότι η οδηγία του 2008 που αφορά τους υφισταμένους και τη θέση τους σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας ισχύει ήδη στις θαλάσσιες μεταφορές για τους ναυτικούς και τους αλείς. Η 24 αφαιρεί κάθε δυνατότητα εξαίρεση στις συλλογικές απολύσεις και οι εθνικές διατάξεις για τις συλλογικές απολύσεις που ισχύουν σε πολλά κράτη-μέλη αντικατοπτρίζουν τα ίδιο χαρακτηριστικά των θαλάσσιων ε, μεταφορών. Άρα τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να ορίζουν αν χρειάζονται νέα νομοθετικά μέτρα και σε περίπτωση κατάφασης θα προβάλλουν προτάσεις που να αντικατοπτρίζουν πραγματικά τις απαιτήσεις του θαλάσσιου τομέα μεταφορών. Άρα η αρχική μου πρόταση επιτρέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης ορίζοντας όρια. Η 30 όπου ζητάμε μείωση από 5 σε 2 χρόνια την θέση ισχύ αυτής της οδηγίας ε, θεωρώ ότι ο χρόνος είναι ανεπαρκής. Ιδιαίτερα επειδή θα πρέπει να επέλθουν αλλαγές σε 8 κράτη-μέλη. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς προς αυτούς. Δεν μπορούμε να ε, θέσουμε σε ισχύ αυτή την οδηγία σε δύο χρόνια σε 28 κράτη-μέλη. Αυτό είναι καθαρή ουτοπία. Δεν αντιτίθεμαι, μακάρι να μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο σε δύο χρόνια. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο. Χρειάζονται πέντε χρόνια, θεωρώ, πριν από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας. Ως προς τελευταία τροπολογία δεν, δεν διαφωνώ ως προς την ουσία, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές. Δεν θα μπορούσαμε σε δύο χρόνια να εφαρμόσουμε αυτή την οδηγία. Και μετά μπαίνουμε σε διαδικασία παράβασης που είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας. Ελπίζω να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους συναδέλφους μέχρι τον Απρίλιο. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο ε, στην σκιώδη συγγήτρια του SND Παλτατσίνο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μόλις ενημερώθηκα από την εισηγήτρια ότι για το πρώτο μέρος και λυπάμαι που δεν ήμουν να παρούσα, άργησα. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ στις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει διότι η πρόταση της Κομισιόν σαφώς έχει στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες των ναυτικών. Με τις δικές μας τροπολογίες θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι θα έχουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας οι ναυτικοί. Θα πρέπει να έχουν δίκαιες συνθήκες απασχόλησης και κοινωνική προστασία. Να είμαι απόλυτα σαφής λοιπόν. Δεν σκοπεύω να μπλοκάρω καμία πώληση πλοίων, αλλά με τις τροπολογίες μας επιτρέπουμε κάποιες παρεκκλήσεις, αλλά με τη συμφωνία όλων των ενδιαφερομένων. Δηλαδή, των ε, δημοσίων αρχών, των εργοδοτών και των εργαζομένων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες του τομέα αυτού. Θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται αυτές ενώ θέλουμε να βελτιώσουμε και τα αποτελέσματα της εργασίας. Η Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας έχει δείξει πώς μπορεί να υπάρξει ένας κοινός δρόμος Γι' αυτό η σύμβαση αυτή αποτέλεσε σαφω βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τρεις βασικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει μία σύμβαση η οποία σαφώς έχει στόχο να βελτιώσει τα δικαιώματα των εργαζομένων σε διεθνέ επίπεδο. Δεύτερον, τα δικαιώματα των ναυτικών έχουν βελτιωθεί, υπάρχουν καλύτερα εχέγγυα. Τρίτον, η οδηγία εφαρμόζει μια συμφωνία ανάμεσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών ε, και τους ε, εφοπλιστές. Η συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων έχει μεγάλη συμφωνία τη βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τα, οι τροπολογίες που προτείνονται από τη δική μας πλευρά καλύπτουν τομείς που δεν ρυθμίζονται από τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίζουμε να μην υπάρχει προτιμησιακή μεταχείριση κάποιων σκαφών στα ίδια ύδατα. Γι' αυτό υποβάλλουμε τροπολογία ώστε να είμαστε βεβαίοι ότι τα σκάφη που δεν είναι ενιολογημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που όμως πλέουν σε ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, δεν ε, θα έχουν καλύτερη μεταχείριση. Θα πρέπει λοιπόν ε, να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων εφόσον βρίσκεται σε ε, εδαφικά έδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσχετα από, το που, ε, άσχετα από τη σημαία που έχει το σκάφος. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με όλες τις τεχνολογικές ε, βελτιώσεις ε, μπορεί να υπάρχει διαβούλευση με τους εργαζομένους, ακόμα και όταν βρίσκονται στις ανοιχτές θάλασσες. Η θέση μας είναι ότι οι ναυτικοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες και θα πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα να συζητούν τη θέση τους ε, με τους εργοδότες. Αυτό είναι βασικός τρόπος για να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών. Επίσης προτείνουμε να υπάρχει δυνατότητα διαλόγου και συμφωνίας σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων. Η Κομισιόν προτείνει αποκλήσεις εφόσον υπάρξει διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων. Αλλά αποκλεισμό των δικαιωμάτων αυτών θα σημαίνει ότι οι ναυτικοί θα βρεθούν χωρί ε, θέση απασχόλησης και δεν θα μπορούν να υψώσουν τη φωνή του ε, όσον αφορά αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τους ε, εργοδότες τους. Μπορεί λοιπόν να αντιμετωπίσουν αποφάσεις οι οποίες μπορούν να αποφευθούν ε, με τη σωστή διαβούλευση. Η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων ε, ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το νομοθέτημα και μία κατηγορία εργαζομένων που είχαν ελάχιστη ή καμία προστασία λαμβάνουν τώρα νέα δικαιώματα. Είναι καθήκον μας απέναντι σε αυτούς τους εργαζομένους. Δεν μπορούμε να να κλείσουμε τα μάτια και να αφήσουμε όσοι έχουν τις συνθήκες των εργαζομένων αυτών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα. Οι τροπολογίες αυτές ε, θα σταθεροποιήσουν περαιτέρω τα δικαίματα αυτά. Ε, και στο μεταξύ η οδηγία αυτή δεν είναι καθόλου καινοτόμα όσον αφορά τον αριθμό των ετών διότι υπάρχει ήδη σύστημα. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί απέναντι σε περαιτέρω συζητήσεις και πολύ ευχαριστώ. Ε, θα ανταποκριθούμε σε προσκλήσεις για να βρεθεί μια κοινή λύση στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω εκ μέλους του συναδέλφου Φιλίντε Μπάκεμ δεν κατέθεσε τροπολογίε από αυτού του φακέλου. Ανέφερε κατά τη διάρκεια της τελευταίας συζήτηση ε, ότι θεωρεί ότι η συγγήτρια έκανε μία καλή πρόταση και βρήκε την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ της ε, ελκυστικότητας του κλάδου αλλά και της ιδιαίτερη κατάστασης ε, αυτού του κλάδου που καθιστά δύσκολη την εφαρμογή όλης της κοινωνικής νομοθεσίας σε αυτό το τομέα. Αναγνωρίζει λοιπόν την ανάγκη για μια καλή προστασία των ναυτικών, αλλά και την ιδιαίτερη κατάσταση ε, σε ό,τι αφορά την εργασία ε, εντό ενός σκάφου. Πρέπει να γίνει και μια αναφορά στην ναυτιλία. ο τομέα είναι πολύ ανταγωνιστικό ε, και οι πλειοκτήτε, οι εφοπλιστέ πολύ εύκολα μπορούν να αλλάξουν σημαία και να πάρουν μια σημαία μη του μέλου. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες με τις οποίες δεν συμφωνεί, που διατηρούν το 2023 της Επιτροπής για τη μεταφορά των επιχειρήσεων ε, του πεδίου εφαρμογή θεωρεί ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η οδηγία αυτή μπορεί να προωθεί στην προστασία, την κοινωνική προστασία των εργαζομένων, αλλά μόνο ε, την προστασία κάποιων ε, εργοστασίων, για παράδειγμα, όχι στα κινητά αγαθά εφόσον εργαζόμενοι εδώ εργάζονται ε, σε ένα σκάφος, σημαίνει ότι βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση. Μετά για τις ε, πληροφορίες ε, και τις διαβουλεύσεις θεωρείται ότι, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει εξαίρεση για τους ναυτικούς. Συμφωνεί λοιπόν εδώ με την πρόταση της Επιτροπής και της Τροπολογίας της Συγήτριας και το ίδιο ισχύει για την 98 κάθετος 59 της Επιτροπής όπου θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις και πάλι για τους ναυτικούς. Καθώς ε, η απασχόληση ε, είναι περίπλοκη, θα δώσει αυτή η οδηγία κίνητρο στους πλειοκτήτες να αλλάξουν τις πρακτικές τους. Ε, ο κύριος Δεμπάκε θέλει να ε, καταλήξουμε σε ε, καλούς συμβασμούς για να στηρίξουμε τον τομέα της ναυτιλίας ε, που είναι σημαντικό τμήμα της οικονομίας και σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία. Θέλει πως η Επιτροπή να παρέμβει, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. σε ό,τι αφορά τι προτάσει, ε, τι τροπολογίε που επιβλήθησαν και τη σημερινή συζήτηση δείχνουν ε, την ισχυρή δέσμευση κάποιων αξιότιμων μελών του Κοινοβουλίου για τη συμπερίληψη των ε, ναυτικών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οδηγιών περί απασχόλησης. Ίσως όμως θα θέλαμε να διευκρινίσουμε κάποια στοιχεία που θα βοηθήσουν τη συζήτηση. Σε ό,τι αφορά τι τροπολογιε 20 και 21, η οδηγία περιφερειακότητας εξαιρεί τους αλληλείς και ε, άλλες και άλλε κατηγορίε εργαζομένων. Προτείνεται εδώ να συμπεριληφθούν ε, στην ε, οδηγία φερεγγιότητα. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους σε κατοικίε, θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάστασή τους. Εμείς δράσαμε ενεργά στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του ILO για αυτό το ζήτημα και έχουν αντιδοτηθεί τα κρατημέλη να κυρώσουν αυτή την πολύ σημαντική σύμβαση. Όμως η συμπερίληψη αυτών των εργαζομένων δεν συμπεριλήφθη ε, στην αξιολόγηση αντικτύπου για αυτή την πρόταση. Για τις τροπολογίες 24-29 και για τις απολύσεις και για την μεταφορά των επιχειρήσεων και αυτές τις δύο οδηγίες θεωρούμε ότι ε, η δεν θέλουμε να έχουμε πολύ μεγάλο κόστος ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να λάβουμε υπόψη την, ε, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτού του κλάδου με, την, με τις αγοραπολισίες καφών. Για την τροπολογία 27, βάσει των υφιστάμενων αρχών ναυτιλία, όπως η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της θάλασσα, το... Ε, η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά τα σκάφη που είναι καταχωρισμένα, νιολογημένα σε κράτη-μέλη. Αυτό αφορά όλη την νομοθεσία ε, και έτσι δεν μπορεί να ισχύσει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκάφη που, είναι, που πλέουν ε, υπό παναμική σημαία και πλέουν στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν μια μεταβατική περίοδος 5 ετών. Προτάθηκε να, για να ληφθεί υπόψη η διαφορετική κατάσταση που υπάρχει στα κρατημέλη τα κράτη-μέλη δεν αξιοποιούν αυτές τις εξαιρέσεις ε, στον ίδιο βαθμό. Κάποιες ε, εξαιρούν τους ναυτικού, κάποια κράτη-μέλη εξαιρούν τους ναυτικούς μόνο από τη μία ε, οδηγία, ενώ κάποια άλλη από όλε. Γι' αυτό θα προτείνουμε αυτή την πενταετή περίοδο. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε το λόγο και πάλι στην εισηγήτρια. Ειλικρινά δεν έχω πολλά να προσθέσω σε σχέση με αυτά που είπα πριν. Μόνο δύο στοιχεία ως προς το διαδίκτυο. Δηλαδή το θέμα που σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες. Επαναλαμβάνω αυτό που προείπα. Όταν εμείς ως νομοθέτες ε, καλούμαστε να δημιουργήσουμε, να νομοθετήσουμε και ε, καθόμαστε ε, σε ένα έδρανο και ορίζουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο του μέλλοντος, θα πρέπει να πατάμε με τα πόδια μας στη γη. Γιατί να προτείνουμε ένα νόμο ε, χωρίς να έχουμε του, τους σπόρους τότε θα παραμείνει νεκρό οράμα. Δηλαδή, ας προχωρήσουμε με αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Το διαδίκτυο είναι δαπανηρό, είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Θα χρειαζόταν μία μελέτη που γίνονται πολλές αναδιαστήματα, άλλες είναι χρήσιμες, άλλες όχι. Και χρειάζεται ειδική νομοθέτηση για την προστασία η ναυτική εκεί προστατεύονται από τις εθνικές νομοθεσίες. Γιατί να περνάμε ένα μήνυμα ότι δεν προστατεύονται, τότε δημιουργεί λάθος εντυπώσεις. Ε, σωστός ο εξυγχρονισμός, αλλά να ε, λάβουμε υπόψη και τις γραφειοκρατικές ή διοικητικές δαπάνες που πλήττουν όλους τους φορείς και τους επιχειρηματίες και ιδιαίτερα ε, αυτόν τον τομέα. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ε, επιπρόσθετες δαπάνες ε, για έναν τόσο ευάλωτο τομέα. Όλοι οι συνδικάτα, εφοπλιστές, ναυτικοί, εργαζόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικών απολύσεων. Η διαβούλευση όμως δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική και δεσμευτική. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή αντιπαράθεση, αλλά δεν θα πρέπει ο καθένας να, να κλείνεται στο, στο δικό του κέλυφος και να μην λαμβάνει υπόψη τους ε, υπόλοιπους. Δεν θέλω να απαντήσω στην Επιτροπή γιατί θα γίνω πολύ κακιά και σταματάω εδώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών στις 18 ε, Μαρτίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Απασχόλησης στις 18 Μαρτίου, ίσως ε, τον Απρίλιο στην Ολομέλεια, κατά τη δεύτερη Ολομέλεια, τη δεύτερη σύνοδο. Μπορούμε να επανέλθουμε στο σημείο 14, διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην κοινότητα. Η Επιτροπή Απασχόλησης υιοθέτησε την έκθεση και μπορώ να δώσω το λόγο στην ε, εισηγήτρια την κυρία Στανόκα. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματοποιήθηκε ο τριμερής διάλογος και όπως ανέφερα το Δεκέμβριο η απόφαση της Κορεπέρ δεν ικανοποίησε το Κοινοβούλιο. Δεν μπορέσαμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας πέρσι. Η νέα ελληνική Προεδρία τον Ιανουάριο υπέβαλε συμβαστικές προτάσεις. Η συμφωνία αυτή έχει να κάνει με τα μοντέλα ad hoc και η θέση του Κοινοβουλίου είναι ότι πρέπει να έχουμε λέγει όσον αφορά το μέγεθος του δείγματος καθώς και άλλα χαρακτηριστικά τέτοιων μοντέλων ad hoc καθότι είναι πολιτικό ζήτημα το πώς θα καθορίζονται οι έρευνες αυτές που θα πραγματοποιούνται μία φορά το χρόνο και που θα είναι αφιερωμένες σε ιδιαίτερες μελέτες, θα αφορούν ιδιαίτερα ζητήματα όπως είναι η ανεργία των νέων, οι συνθήκες απασχόλησης των μεταναστών κλπ. κλπ. Τώρα λοιπόν έχουμε συζητήσει τις προτάσεις ε, της Ελληνικής Προεδρίας. Προτείνονται εδώ κάποια επιμέρους μοντέλα. Μερική χρήση κατευθυνότηση πράξεων και μερική χρήση εκτελεστικών πράξεων για τον καθορισμό αυτών. Και η διαπραγματευτική ομάδα έδωσε εντολή στη γραμματεία μας και τη νομική υπηρεσία μας, ώστε να συζητήσουν να πραγματοποιήσουν μια τεχνική συνάντηση για να συζητήσουν περαιτέρω τι θα αποτελεί αντικείμενο κατεξοδότηση πράξης και τι εκτελεστικής πράξης. Είμαι ε, ευγνώμων ε, προς την πρόεδρό μας ε, που διεύθυνε τις συναντήσεις αυτές και φυσικά είμαι ευγνώμων και προς τη γραμματεία που είναι διατεθειμένη να αναλάβει το θέμα αυτό για να πραγματοποιηθούν οι συζητήσεις με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εάν βρεθεί μια λύση την οποία να μπορεί να ε, δεχθεί η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης 18 Μαρτίου το αργότερο. Αυτό ήταν το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα, διότι Μετά την ψηφοφορία θα συζητήσουμε το σημείο 16 γύρω στις 11.30. Καλό βράδυ.